Ε, συνεπές με τις μεγάλες πολιτικές και προσεγγίσεις που ε, υποστήριξε από την αρχή της εκδήλωσης της κρίσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η ε, συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο θέμα μας είναι συζήτηση επί της εκθέσεως του David Μάρτιν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη άσκηση του δικαιώματο εξέταση των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δίδω το λόγο στον κύριο Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, κάποιες ευχαριστίες. Στην γραμματεία της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων και τον Τόμας ε, Κάσκι για την ε, βοήθεια που μας έδωσε στη σύνταξη της έκθεσης. Ευχαριστώ και τον ε, Πίτροπο Σεύκοβιτσε και τη Δανική Προεδρία, διότι πολύ νωρίς εντάχθηκαν στη διαδικασία αυτή. Η συμβολή του στην Επιτροπή ΑΦΚΟ και προς εμένα προσωπικά ήταν πολύ ευπρόσδεκτη και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία μαζί τους για να φτάσουμε σε μια ικανοποιητική συμφωνία για όλα τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ επίσης τους κοιόδης των άλλων πολιτικών ομάδων για την πολύ ε, μεγάλη συνεργασία στα πλαίσια της οποίας διαπραγματευτήκαμε την έκθεση. Είναι φιλόδοξη η έκθεση αυτή και πολύ επίκαιρη επίσης μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Το 1995 ήμουν εισηγητής του Κοινοβουλίου για τη συνθήκη του Μάστριχτ και επιτυχώς ζητήσαμε να αναβαθμίσουμε την δυνατότητα του Κοινοβουλίου ε, για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών ε, συμπεριλαμβάνοντας το δικαίωμα αυτό στη συνθήκη. Από τότε δεν έγιναν αλλαγές οι τροποποιήσεις. Υπάρχει δυνατότητα ε, να αντιμετωπίζει με εξεταστικές επιτροπές στο Κοινοβούλιο καταγγελίες για κακοδιοίκηση ή παραβιάσεις. Οι επιτροπές μπορούν να απευθύνονται σε ενεχόμενα άτομα για να διαπιστώνουν αν υπήρξαν παραβάσεις του δικαίου ή προβλήματα ε, διαφθοράς ε, στην ε, εφαρμογή του δικαίου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντική η άσκηση αυτή ως αρχή. Το λέω αυτό πριν μπω στη διαδικασία και στην ουσία της έκθεσης. Υπήρξαν στην ιστορία του Κοινοβουλίου τρει εξεταστικέ επιτροπέ, η μία για το καθεστώ διαμετακόμιση, η άλλη για τη σπογγόδη κεφαλοπάθεια και πρόσφατα για την Equitable Life, την ασφαλιστική εταιρεία. Η εξεταστική αυτή η τελευταία ε, οδήγησε ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα να φτάσει στην αλήθεια, γιατί δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε με του ενδιαφερομένου, δεν μπορούσαμε να διασφαλίσουμε πρόσβαση στα έγγραφα και δεν υπήρχαν ε, επιπτώσει αν κάποιο ε, έκανε ψευδεί καταθέσει. Η τελευταία λοιπόν επιτροπή έδωσε μεγάλη μάχη για να αποκαλύψει την αλήθεια. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες απέκτησε πολλά προνόμια και αναβαθμίστηκε το Κοινοβούλιο. Έπρεπε όμω και το ζήτημα αυτό να προσαρμοστεί στι ανάγκε του 21ου αιώνα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ε, ε, ε λάβουμε υπόψη μα ότι ενώ αναβαθμιστήκαμε σε πολλά άλλα θέματα, σε θέματα ε, εξεταστικών επιτροπών δεν είχαμε αναβαθμιστεί. Έπρεπε λοιπόν να ισχυροποιηθούμε. Ε, η ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να εξετάζει θέματα κακοδιοίκηση ευρωπαϊκού δικαίου για λογαριασμό των Ευρωπαίων πολιτών, όπω γίνεται και στο εθνικό επίπεδο ανάλογα για, το εθνικό, για τα εθνικά κράτη και τι διοικήσει. Ε, όπω είπε ο μεγάλο φιλόσοφο Μπομπ Ντίλαν, ε, η, αλήθεια είναι βέλο και στενή πύλη που διαπερνά. Ε, έτσι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια για να δούμε το παρελθόν. Χρειάζεται πρόσβαση σε έγγραφα, επαφή με πρόσωπα. Αλλιώ δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να είναι αποτελεσματικό στο δημοκρατικό του καθήκον. Αυτό είναι ένα ε, ρόλο που τον αναλαμβάνει ε, χωρί επιπολαιότητε αλλά με κάθε σοβαρότητα το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να μην υπάρχει φόβος ότι θα γίνει κατάχρηση του, ε, της δυνατότητας αυτής. Γιατί γίνεται η μεταρρύθμιση τώρα. Πρώτον, διότι πάρα πολλά θέματα εκκρεμούσαν μετά την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής για την Equitable Life και τις συστάσεις που έκανε και επειδή η συνθήκη της Λισαβόνας αναβάθμισε σε ε, κανονισμό το θέμα των εξεταστικών επιτροπών και μάλιστα με βάση το άρθρο 226 συνθήκης ε, ε, το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει πρωτοβουλία για μια πολιτική. Εδώ ε, βέβαια ε, μπορούμε να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες αλλά που θα πρέπει να εγκρίνονται από τα άλλα δύο ε, θεσμικά όργανα. Πρόεδρε, νόμιζα ότι είχα έξι λεπτά. Αν, αν τα μοιράσετε... Όχι, θα ήθελα να κάνω την παρουσίαση ολόκληρη της έκθεσης τώρα. Γιατί τώρα πάνω από στην ουσία. Είναι σημαντικό αυτό. τώρα να το πω, όχι στο τέλος. Υπάρχουν λοιπόν τρία ε, σημαντικά στοιχεία ε, που αναφέρω για τις εξεταστικές επιτροπές. Πρώτον, η δυνατότητα να απευθύνεται άμεσα στα ενεχόμενα πρόσωπα στο θέμα. Ένα μείζον θέμα, το οποίο το είδαμε από την εξεταστική στην Equitable Life, ήταν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να ε, ζητήσουμε, να εξετάσουμε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πολλές φορές έστελναν αντιπρόσωπο κάποια θεσμικά όργανα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που ελήφθησαν για να απευθυνόμεθα άμεσα στους ενεχομένους ή στους εμπειρογνώμονες σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι η στους εμπειρογνωμονες σε καποιο συγκεκριμενο θεμα ενα δευτερο θεμα ειναι η πρόσβαση στα έγγραφα και η δυνατότητα της Επιτροπής να εξετάζει έγγραφα που έχουν άμεση σχέση με την εξετάση ε, την έρευνα. Επίσης η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζεται και να βλέπει επιτόπου το πλαίσιο της έρευνας. Από παλιές έρευνες ξέρουμε ότι οποιαδήποτε μορφή κύρωσης για άρνηση κατάθεσης ή δωροδοκία ή ψευδορκία ε, ε, δεν υπήρχαν κυρώσει. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει την ίδια βάση για κυρώσει όπω αυτέ που υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη. Η έκθεσή μου καταρτίστηκε και στηρίχθηκε σε πολύ λεπτομερεί εκθέσει Εθνικών Κοινοβουλίων για τι Εξεταστικέ Επιτροπέ. Βεβαίω το Κοινοβούλιο δεν είναι δικαστήριο. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, κυρώσεις ε, για ψευδορικία κλπ. Αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη και συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει στα πλαίσια της μεταρρύθμισης αυτής. Όμως, σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα, η εντολή της Εξεταστικής Επιτροπής είναι απλή η αποκάλυψη της αλήθειας. Δεν ε, επιβάλλουμε κυρώσεις, δεν αναλαμβάνουμε νομική δράση. Αυτό ε, είναι συστάσεις, ε, αυτά περιλαμβάνονται στις συστάσεις που θα κάνουμε. Ελπίζω να ολοκληρωθεί θετικά η έκθεση αυτή και είμαι αισιόδοξο ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να καταλήξουν στη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα δώσω το λόγο στο Συμβούλιο των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον κύριο Νικολάη Βάμεν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι βουλευτές, κύριε τη Πρόεδρε της Επιτροπής, το δικαίωμα ερεύνης είναι ένα απόλυτο δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εποπτικών εξουσιών του επιτρέπει στην Εξεταστική Επιτροπή να διερευνήσει ε, καταγγελίες περί ε, αντικανονικότητας ή ατασταλιών. Η συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε καινούργιες διατάξεις όσον αφορά την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Οι διατάξεις αυτές τώρα καθορίζονται από το Κοινοβούλιο που ενεργεί με τα αποδική του πρωτοβουλία αφού έχει την συνένεση του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Η Προεδρία σέβεται απολύτως το δικαίωμα εξέτασης ε, του Κοινοβουλίου και γι' αυτό και παρακολουθεί στενά, την, παρακολούθησε μάλλον στενά τις εργασίες του κ. Μάρτιν επί της εκθέσεως αυτής. Παρομοίως η Προεδρία εργάστηκε σκληρά εντός του Συμβουλίου ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε επίσημες τριμερείς διαπραγματεύσεις ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων που είχαμε σε αυτό το θέμα με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων τον Ιανουάριο, Υπέδειξε ότι καθώς προέρχομαι από μια χώρα όπου ισχύει η παράδοση διαφάνειας καθώς και έντονου κοινοβουλευτικού ελέγχου θα προσεγγίσουμε το θέμα με ανοιχτό μυαλό και με τη βούληση να βρεθεί κάποια λογική συμβιβαστική λύση. Οι διαπραγματεύσει, οι επαφέ που υπήρξαν ανάμεσα στον εισηγητή και στον Συμβούλιο μετά από την ψηφοφορία στην ΑΦΚΟ επί τη εκθέσεω Μάρτιν ε, παρήχαν μια εξαίρετη ευκαιρία ώστε να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα και να βελτιώσουμε την κατανόηση ε, αλλήλων για το θέμα. Γι' αυτό και θα ήθελα να πω στον κύριο, μάλλον να συγχαρώ τον κύριο Μάρτιν για την ε, ανοιχτή του ε, διάθεση και τον επικοδομητικό διάλογο στον οποίο προσήλθε με την Προεδρία. Δεν υπάρχει λόγος να κρύβουμε το γεγονός ότι το θέμα αυτό είναι πολύ λεπτό για όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα. Ωστόσο, είμαι πεπισμένος ότι ε, οι επαφές που, είχε η Προεδρία με τον κύριο Μάρτιν θα προμηθεύσουν μια καλή βάση για περαιτέρω διοργανικές επαφές. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες περί της ε, έκθεσης, θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία που είναι ιδιαίτερη σημασία για το Συμβούλιο. Καταρχήν, Πιστεύει το Συμβούλιο ότι η θεμελιώδης πολιτική φύση του δικαιώματος εξέταση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να γίνει αποδεκτή εξ αρχής ε, σε σχέση με τους κανόνες έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διάρκεια των, της διαδικασίας. Επίσης, ε, σημαίνει ότι η Επιτροπή αυτή κάθε φορά έχει σχεδόν νομικές αποφάσεις, ε, ε, δικαιοδοσίες μάλλον. Το ίδιο συμβαίνει ότι Μάλλον, θα πρέπει οι εξεταστικές επιτροπές να αποφύγουν κάθε επικάλυψη με αρμοδιότητες άλλων, κρατώ, άλλων κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης κατά τη διάρκεια της άσκησης ε, των αρμοδιοτήτων της. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, εγώ προσβλέπω σε περαιτέρω επαφές με τον κύριο Μάρτιν και την διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου από αυτού του θέματος και θα σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία θα κάνει κάθε τι δυνατό ώστε να επιτευχθεί συμβιβασμό που θα είναι αποδεκτός για τα τρία θεσμικά όργανα και θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να ασκήσει το δικαίωμα εξέτασής του με όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί κύριοι βουλευτέ, στη συνθήκη τη Λισαβόνα συμπεριλαμβάνονταν διάφορε καινοτομίε για το Ευρωκοινοβούλιο. μία από τι καινοτομίε ήταν ακριβώ η, ε, η σύσταση, το δικαίωμα μάλλον σύσταση εξεταστική επιτροπή. Και όλοι θα πρέπει αυτό να το χειροκροτήσουμε. Και τώρα είναι η κοινή μα ευθύνη να εφαρμόσουμε αυτή τη νέα διάταξη όσο γίνεται πιο σύντομα, σε, με επικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα με κοινή λογική και με πλήρη σεβασμό στο άρθρο 226 της Συνθήκης περί λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν ανέκαθεν υποστήριζε την ανάγκη για ισχυρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γι' αυτό και πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις για το σχέδιο του έκθεσης του κ. Μάρτιν και εκτιμώ ιδιαίτερα το πνεύμα συνεργασίας και την καλή συνεργασία που υπήρξε με την Προεδρία και τον ε, Υπουργό Φάμεν. Ήδη ξέραμε από τότε κάποιες ε, από τις προβληματικές σημαντικέ πτυχέ του αρχικού σχεδίου, αλλά μόνο λίγε από τι ανησυχίε μα αντιπροσωπεύονται στο αποτέλεσμα στην τελική διατύπωση δηλαδή τη έκθεση από την ε, ε, Συνταγματική Επιτροπή. Γι' αυτό και η Ουγγρική και τώρα η Δανική Προεδρία εκφράζουν κάποιε ανησυχίε και γι' αυτό και είναι ευπρόσδεκτη η επιθυμία του εισηγητή να λάβει υπόψη κάποιε από αυτέ τι αντιρρήσει. Είμαστε ε, πολύ θετικοί απέναντι στι συμβαστικέ τροπολογίε που υπέβαλε ο κ. Μάρτιν και προσπαθούμε να καλύψουμε κάποιε από τι βασικέ ανησυχίε του Συμβουλίου και τη Επιτροπή. Αλλά μάλλον δεν είναι μυστικό ότι ακόμα πρέπει να συζητηθούν κάποια στοιχεία πριν να δώσει την απαραίτητη συνένεση που προβλέπεται από το άρθρο 226 η Κομισιόν. Να, υποστη... να τονίσω κάποια σημαντικά στοιχεία για την Κομισιόν. Πιστεύουμε ότι το πεδίο εφαρμογή του μελλοντικού κανονισμού θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο όπω την ε, σημερινή απόφαση. Όπω δηλώνει το άρθρο 226, το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να συστήσει εξεταστική επιτροπή στην άσκηση των καθηκόντων του με βάση το άρθρο 13 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι περιορισμοί που αναφέρονται στην ίδια τη συνθήκη. Εμείς ε, καλωσορίζουμε λοιπόν τις συμβαστικές αστροπολογίες ως προς αυτό το στοιχείο. Δεν θα, πρέπει επίσης να καταγράψουμε ότι οι αλλαγές στο άρθρο 226 αφορούν τη διαδικασία και όχι το αντικείμενο των εξεταστικών επιτροπών που είναι βασικά πολιτικό εργαλείο και όχι νομικό στη διάθεση του Κοινοβουλίου για την άσκηση του πολιτικού ελέγχου. Γι' αυτό και πιστεύω περαιτέρω συζήτηση θα χρειαστεί για τα διερευνητικά εργαλεία που προτείνονται στο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που φαίνονται να είναι υπερβολικά. Τέλο, θα ήθελα επίση να αναφέρω το άρθρο 17 του σχεδίου κανονισμού που αφορά την ακρόαση υπαλλήλων και άλλων λειτουργών της Ένωσης και των κρατών μελών. Οι συμβαστικές τροπολογίες αντιμετωπίζουν μάλλον κάποιες από τις βασικές μας ανησυχίες όσον αφορά την ελευθερία ε, ε, μαρτυρίας και επίσης ε, τα συμπεράσματα αλλά παραμένει κάποια απορία όσον αφορά τη διαφορετική μεταχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών υπαλλήλων που δεν αιτιολογείται αντικειμενικά. Η Κομισιόν επίσης καλωσορίζει την ε, πρόθεσή σας να κάνετε κάποιες τροπολογίες για την έκθεσή σας, αλλά όχι για το νομοθετικό ψήφισμα, γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα να, στα τρία όργανα να προβούν σε επικοδομητικές τριμερείς συζητήσεις έτσι ώστε το Συμβούλιο και οι Κομισιόν να μπορέσουν εύκολα να δώσουν τη συνένεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 226 αφού το Κοινοβούλιο θα έχει ψηφίσει επί του νομοθετικού ψηφίσματος. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία μαζί σα και με το Συμβούλιο ώστε να επιτύχουμε έγκαιρη και επιτυχή έκβαση για αυτό το σημαντικό φάκελο. Ευχαριστώ. Και τώρα ακολουθούν οι μιλητέ. Πρώτο ο κύριο Βίλαντ. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ένα όργανο που είναι αρμόδιο για ε, την παραγωγή της νομοθεσίας θα πρέπει να είναι αρμόδιο και για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν αφορά μόνο λοιπόν, το κοινοτικό κεκτημένο αλλά και την εφαρμογή και την υλοποίηση του κοινοτικού δικαίου. Και είναι πολλά τα στρεβλά ε, είδαμε και από την Εξεταστική Επιτροπή για το Equitable Life. Ε, είναι πολύ αξιοπερίεργα αυτά που προέκυψαν ως προς τα πραγματικά περιστατικά αλλά και η συνέχεια ε, που δόθηκε θα πρέπει να μην σταματήσει εδώ. Θα ήθελα να σας αναφέρω τα σημαντικότερα σημεία για την ομάδα μου. Πρώτον, καταλαβαίνουμε ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν επιφυλάξεις εάν ε, υπάρχει εύλογος λόγος ε, να μην ε, καταθέτουν υπουργοί και υπάλληλοι. Αλλά η απόφαση δεν θα πρέπει να είναι αυθαίρετη, αλλά δικαιολογημένη και τεκμηριωμένη. Δεύτερον, δεν μπορεί να είναι στη διακριτική ευχαίρεια του μάρτυρα αν θα είναι δημόσια κρόση και κλεισμένο των θυρών. Τρίτον, ο κάθε μάρτυρα θα πρέπει προφανώ να λέγει την αλήθεια. Τέταρτον, αναμένουμε από τα κράτη-μέλη, εκείνοι που δεν λέγουν την αλήθεια, τουλάχιστον να τιμωρούνται όπω τιμωρούνται εκείνοι που ψευδομαρτυρούν ε, στα αρμόδια εθνικά όργανα. Πέμπτον, αυτό αφορά την τροπολογία 31, ε, ε, για την ομάδα μας είναι σημαντικό στο τέλος ε, των εργασιών μιας εξεταστικής επιτροπής να υπάρχει και ψήφος μειοψηφίες. Λυπάμαι που δεν θεωρήθηκε παραδεκτή αυτή η τροπολογία από τον πρόεδρο ή τις υπηρεσίες του, το θεωρώ λάθος. Τέλος, και το Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασαν ικανοποίηση και χαρά για την προθυμία του Κοινοβουλίου σε συμβιβασμό. Εγώ θα χαιρόμουν αν τελικά αυτή η χαρά για την προθυμία συμβασμού ε, δεν ήταν μονόδρομος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γκουαλτιέρη, παρακαλώ. Πόρτο Μάρτιν, η έκθεση Μάρτιν ανοίγει το δρόμο για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης που ορίζουν ε, το δικαίωμα εξέτασης Πρόκειται για μια θεμελιώδη λειτουργία του Κοινοβουλίου, τη λειτουργία του πολιτικού ελέγχου. Η συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει μια ε, συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία και γι' αυτό και ευχόμεθα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, Συμβούλιο και Κομισιόν να φτάσουν στο πνεύμα αυτού του κανόνα που αναθέτει το ρόλο της εξέτασης στο ίδιο το Κοινοβούλιο και περιορίζει το ρόλο του, Συμβουλίου και της Κομισιόν σε μια συνένεση. Ο εισηγητής Μάρτιν ε, χρησιμοποιεί τις προηγούμενες ε, σχετικές εκθέσεις. Αυτό το μέσο σημαίνει συγκεκριμένα όρια και συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Η Ουγγρική και η Ιδανική και η Προεδρία έχουν ε, προτείνει κάποιες ικανοποιητικές συμβαστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στα αιτήματα της Κομισιόν και κάποιων κρατών μελών, αλλά δεν περιορίζουν το δικαίωμα του Κοινοβουλίου για τη σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και για τον εντοπισμό της ε, κακοδιαχείρισης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινίσουμε κάποιες διατυπώσεις. Είναι σημαντικό να μην ε, κάνουμε πίσω σε ένα σημείο. Οι εξεταστικέ επιτροπές να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στα έγγραφα και στους, στα άτομα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με νομικές, νομικό έλεγχο, αλλά ακριβώ για την εφαρμογή του πολιτικού δικαιώματος ελέγχου που επικυρώνονται από τη συνθήκη Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Γιάτα Ενμάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή David Μάρτιν για την εξαιρετική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται καλή διακυβέρνηση, δημοκρατική και διαφανή. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα σχετικά έγγραφα, αναφέρθηκε αυτό. Σήμερα σε αυτό το θέμα δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Επιτροπή και Συμβούλιο είναι κατά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ποιες αρμοδιότητες έχει το Κοινοβούλιο εποπτεύοντας τις κυβερνήσεις μέσα από τέτοιες εξεταστικές επιτροπές. Πρόκειται για πολιτικό έλεγχο υπάρχει ο έλεγχος και από τα δικαστήρια και πρέπει να διακρίνουμε με μεταξύ των δύο μορφών ελέγχου. Σε αυτά τα πλαίσια το Κοινοβούλιο χρειάζεται για τον πολιτικό έλεγχο ισχυρές αρμοδιότητες. Μεταξύ άλλων όμως δεν νομίζω ότι συγκαταλέγεται όπως είπε ο Επίτροπος το ότι θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι εθνικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικοί υπάλληλοι απέναντι στο Κοινοβούλιο είναι σε, στην ίδια θέση όπως και η Επίτροπη και πρέπει και εκείνοι να μπορούν να ερωτώνται όπως όλοι οι άλλοι από τις εξεταστικές επιτροπές. Σημαντικός όμως είναι ο κεντρικός ρόλος της εποπτείας των θεσμικών οργάνων, διότι έτσι ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών. Η εμπιστοσύνη αυτή της πράξης μας θα πρέπει να ενισχυθεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο καθήκον και όταν μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις σχετικές μας αρμοδιότητες, τότε σίγουρα θα καταφέρουμε να ε, χρησιμοποιούμε σωστά και όχι συχνά το όργανο αυτό. Ο κύριος Έφνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η δημοκρατία χρειάζεται διαδικασίες και οι διαδικασίες ε, λειτουργούν τόσο καλά όσο καλοί είναι οι κανόνες που τις διέπουν. Εν προκειμένου, όπως έδειξε και η εμπειρία μας από την Equitable Life και την Εξεταστική Επιτροπή, οι κανόνες εδώ δεν επαρκούν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε επιτέλους ένα λειτουργικό σύστημα εξέτασης όταν υπάρχει ε, πρόβλημα, κακοδιοίκηση, σκάνδαλα, αυτά πρέπει να έρχονται στο φως. Όταν υπάρχουν υποψίες πρέπει να αποκαθιστούμε την αλήθεια. Ε, το ίδιο όταν επιχειρείται να ε, αποκριβεί μια κατάσταση προβληματική ή σκάνδαλο. Όλα τα σχετικά έγγραφα πρέπει να μπορούμε να τα βλέπουμε. Όλους τους σχετικούς μάρτυρες και ενεχομένους πρέπει να τους ακούμε και επί τόπου. Ε, αν κάποιος ε, ψευδορκήσει ή αρνηθεί να καταθέσει αυτό πρέπει να συνεπάγεται επιπτώσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που δυστυχώς δεν πρόκειται να ψηφιστεί σήμερα. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η προσπάθεια διαφώτισης και η ετοιμότητα για διαφώτιση της κατάστασης στην Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι πάντα δεδομένη. Πολλές φορές λαμβάνονται υπόψη εθνικά ή κομματικά συμφέροντα. Δεν έχουν όλοι την ίδια βούληση για εξυχνίαση της υπόθεσης ενώ θεωρητικά θα έπρεπε. Πολλές φορές ε, υπάρχουν μειοψηφίες ε, που ε, αρνούνται να συνεργαστούν. Γι' αυτό θα πρέπει και οι απόψεις αυτές να αναφέρονται στις, στα πορίσματα των εξεταστικών επιτροπών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ πολύ. Ο έλεγχος του κοινοβουλευτικού είναι πολύ σημαντικός και η δουλειά μας δεν είναι μόνο να ψηφίζουμε νομοθετήματα, κάτι που το παρακάνουμε θεωρώ, αλλά να διασφαλίσουμε ότι θα δαπανώνται σοφρόνως τα χρήματα των φορολογουμένων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη. Ο προκάτοχός μου στην ε, Διοδυτική Αγγλία ήταν ο Νίλ Πάρις, ε, ήταν πολύ σημαντικός διότι εκείνος ε, ασχολήθηκε με την Εξεταστική Επιτροπή σε μια μεγάλη υπόθεση του 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο που έδειξε πόσο ε, ανεπαρκώς αντιμετώπισε η τελευταία κυβέρνηση των εργατικών την κρίση. Αυτή η μεταρρύθμιση δείχνει πώς πρέπει να γίνεται μια, εξεταστική των πραγμάτων, μια εξέταση των πραγμάτων. Ε, νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει πολλά σωστά πράγματα, αλλά σε ορισμένα σημεία το παρακάνει. Για παράδειγμα, δίνει το δικαίωμα στο Κοινοβούλιο να κλητεύει ε, μάρτυρες και να τιμωρεί εκείνους που αρνούνται. Η συνθήκη δεν του δίνει αυτές τις εξουσίες του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι ε, το παρακάνουμε ε, εδώ. Επίσης, εις ό,τι αφορά τους υπαλλήλου των εθνικών κυβερνήσεων, οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να λογοδοτούν στους, κυβερν και να υλοποιούν τις, τις ε, υπουργικές αποφάσεις. Νομίζω ότι ε, ρισκάρουμε να υπονομεύσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και υπονομεύουμε την λογοδεσία ε, στους υπουργούς, ε, των υπουργών. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ε, επιτείνουμε τη λογοδοσία ε, για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Εδώ πρέπει να επικεντρωθεί το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει δηλαδή οι γραφειοκράτες των Βρυξελών να τεθούν υπό ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο και εποπτεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλο και περισσότερο χάνεται η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, απομακρύνονται από την πολιτική της Ένωσης σε πολλούς τομείς. Και δεν μπορούμε παρά την έκθεση πρωτοβουλία του κυρίου Μάρτιν αυτού του καιρού και υποστηρίζει ρητά και η πολιτική μου ομάδα αυτή την έκθεση πρωτοβουλία. Περί τίνος πρόκειται περί του άρθρου 14 ε, της Συνθήκης της Αβώνας. Ε, έχει το δικαίωμα όσο και το καθήκον ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγχει και αυτό να μεταφραστεί σε περαιτέρω πρακτικά βήματα και δεν συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ότι ακριβώς αυτή η διεύρυνση του δικαιώματος εξέτασης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι κάτι το επιθυμητό. Μα αλλιώς πώς μπορεί και πώς οφείλει το άρθρο 226 να εφαρμοστεί συγκεκριμένα στην πράξη. Αν χρειαστεί τωρινές εξεταστικές επιτροπές θα πρέπει να συστήνονται έτσι ώστε να ε, υποθέσεις ε, και ε, υποτιθέμενες ατασταλίες και προβλήματα. Είναι μια διαδικασία απαραίτητη για τη διαφάνεια και την εξέταση. Βεβαίως, εξεταστικές επιτροπές στην κοινοβουλευτική δημοκρατία καλούνται να καλύψουν ένα σημαντικό ρόλο και έτσι τα κοινοβούλια έχουν τη δυνατότητα με ανεξαρτησία και με αυτοτέλεια να ελέγχουν τα πραγματικά περιστατικά και ε, είναι και συνταγματική τους υποχρέωση ως εκπροσώπων ε, των πολιτών, ανδρών και γυναικών. Ακριβώς στη σημερινή κατάσταση, ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτω απαραίτητο. Τέλο, συμφωνώ με τους συναδέλφους που λέγουν ότι ε, ε, χρειάζεται οπωσδήποτε και οι γνώμες της μειοψηφία να καταγράφονται. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Η εξέταση της εκτελεστικής εξουσίας είναι βασικό στόχος κάθε κοινοβουλίου. Είναι και δικαίωμα του κοινοβουλίου όμως ε, ε, να ελέγχει ε, την κυβέρνησή του. Ε, Βεβαίω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγχει του κοινοτικού υπαλλήλου, από το πιο χαμηλό βαθμό μέχρι το πιο υψηλό βαθμό. Ωστόσο δεν υπάρχει λόγο να διευρυνθεί αυτή η δικαιοδοσία και προ υπαλλήλου των κρατών μελών. Αυτό είναι και θα πρέπει να είναι λειτουργία των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η Εξεταστική Επιτροπή θα μπορεί να κλητεύει ειδικού υπαλλήλου από τα κράτη-μέλη να δίνουν στοιχεία και δικαστικά δικαστική συνδρομή. Θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το δικαίωμα όπως λέει η τροπολογία 18 του εισηγητή, να ε, μην αποκαλύπτουν ε, κάποιες ε, πληροφορίες που θα βλάψει τις έρευνες των δικών τους κρατών μελών. Επιπλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να προστατεύονται από το δίλημα, να έχουν αντιφατικές εντολές για το τι θα πρέπει να αποκαλύπτουν ή να αποκρύπτουν. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τσασκόφσκι. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάρτιν για το εξαιρετικό του έργο και τους σκιώδης. Ε, ε, πολύ περιορισμένε αρμοδιότητε είχαν δοθεί στι εξεταστικέ επιτροπέ υπό το φω τη συνθήκη του Μάστρου και δεν ήταν σύμφωνε με τι επιθυμίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη συνθήκη του Λισαβόνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε τον ε, πολιτικό δημοκρατικό έλεγχο, επιτόπου έρευνες, ε, αίτηση για έγγραφα, ακροάσεις ε, εθνικών και κοινοτικών υπαλλήλων και ναι, κυρώσεις, κυρώσεις και όχι κύριε Φόξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε συμφωνία με τις εθνικές διαδικασίες από τις εθνικές αρχές. Δεν είμαστε δογματικοί. Για παράδειγμα, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων εγκαταλείψαμε τη χρήση γλώσσα που θα έδινε την εντύπωση ότι οι εξεταστικέ επιτροπέ θα λειτουργούσαν ω δικαστήριο. Αναγνωρίζουμε τη, την, τη δυνατότητα άρνηση συγκεκριμένου υπαλλήλου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή από πλευρά του προϊστάμενού του, αλλά θα έπρεπε να έρθει και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν θα έρθει. Εμείς ε, θέλουμε να υποστηρίξουμε τις αρμοδιότητες αυτού του ε, σώματος που είναι αντίστοιχες με το πολιτικό του κύρος. Θα πρέπει αυτή η διαδικασία να στηριχτεί και να επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ζητήσω να ησυχάσετε. Ε, επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή David Μάρτιν για το έργο του και τη Δανική Προεδρία για την ε, προθυμία που έδειξε να προχωρήσουμε στην έκθεση αυτή. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι αρμοδιότητες των κλασικών κοινοβουλίων. Τρεις πολύ συγκεκριμένες νομοθετική δραστηριότητα, δημοσιονομική δραστηριότητα και ελεγκτική δραστηριότητα. Και μια άλλη που είναι πιο συγκεχημένη αλλά πολύ σημαντική να δίνει πολιτικού προσανατολισμού. Μέσω λοιπόν τη λειτουργία του ελέγχου μπορούν τα κοινοβούλια να ελέγχουν και να ε, τιμωρούν ε, τη δράση της διοίκησης και της κυβερνήσης. Απαιτούν ε, να δίνουν λογαριασμούς και τέλος αποδίδουν και πολιτικές ευθύνες αν χρειάζεται με μηχανισμούς πιο ελαφριούς ή πιο βαρύς ανάλογα. Το δικαίωμα ελέγχου συμπεριλαμβάνει λοιπόν και τις εξεταστικές των πραγμάτων επιτροπές. Γι' αυτό αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή διευρύνει τις λειτουργίες και δραστηριότητες του Κοινοβουλίου που προχώρησε πολύ στην νομοθετική πτυχή και στις ε, δημοσιονομικές του εξουσίες αλλά υπολείπεται σε ό,τι αφορά τον έλεγχο. Γι' αυτό επειδή ακόμα ε, έχουμε διαδικασία διαπραγμάτευσης μετά την ψηφοφορία, ζητώ από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τον εισηγητή και το Κοινοβούλιο να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα και της εξεταστικής λειτουργίας. Ευχαριστώ. Κύριος Νταφ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ βέβαια. ότι το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται ούτε επιδιώκει ιονή δικαστικές ε, εξουσίες. Όμως, παρόλα αυτά, χρειάζεται μία υπολογίσιμη αρμοδιότητα στην εξέταση σύνθετων πολιτικών ε, προβλημάτων. Προσβλέπω στη συνέχεια του θέματος γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την άνηση μεταχείριση ε, που αναφέρεται στο σχέδιο ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εθνικούς υπαλλήλους. Παράλληλα όμως θα πρέπει να επιδιώξουμε επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα σωστά ένδικα μέσα. Ε, που θα οδηγήσουν στα συμπεράσματα μιας ε, εξεταστικής επιτροπής. Ευχαριστώ. Αρχίζει η διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Μικολάτσικ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι εξεταστικές αρμοδιότητες συγκαταλέγονται στις αρμοδιότητες όλων των κοινοβουλίων, σε όλον τον κόσμο. Η βασική προϋπόθεση ε, για την αποκατάσταση της αλήθειας είναι το δικαίωμα άσκησης αυτού του δικαιώματος. Υπάρχουν λοιπόν αρμοδιότητες και για το κοινοβουλίο μας από τη συνθήκη της Λισαβόνα. Με τη συνθήκη αυτή ε, ε, επιτείνεται ο δημοκρατικός έλεγχος και το άμεσα εκλεγμένο κοινοβούλιο μπορεί να ε, προβαίνει σε εξεταστικές επιτροπές. Ο κανονισμός Νομίζω ότι είναι σωστό εν ώψη της νέα θέση του Κοινοβουλίου και τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Η συζήτηση θα συνεχιστεί. Παρακαλώ ησυχία. Η κυρία Γκίνε για ένα λεπτό στα πλαίσια τη διαδικασία Catch Σα Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να στηρίξω τα σχόλια του εισηγητή μα και να τον ευχαριστήσω για αυτά. Εγώ μιλώ ω πρόεδρο τη Εξεταστική Επιτροπή για την ε, ισότιμη... για το Equitable Life. Να σας πω ότι ο λόγος για αυτή την Εξεταστική Επιτροπή ήταν ότι πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες ε, μας πίεσαν για να κάνουμε τη δουλειά μα, που την κάναμε. Επίσης, ε, δίνει συνέχεια στι Επιτροπές της Εξεταστικής ακόμα δεν έχουμε αποτέλεσμα μετά από τα δικά μας πορίσματα και θα ήθελα οι Βρετανικές Αρχές αν όλοι οι πολίτε που ε, ζημιώθηκαν θα πληρωθούν και πότε. Δεν θα πρέπει να μιλήσουμε μόνο για τις διαδικασίε που είναι σημαντικές και που στηρίζω τις αλλαγές, αλλά και για τη συνέχεια που δίνεται στη δουλειά των διαφόρων εξεταστικών επιτροπών, γιατί ε, το, θα κριθούμε όχι από την έκθεση, αλλά από τις ενέργειες τις οποίες θα προβούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα για τις τελικές παρατηρήσεις θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Επίτροπο Σεύκοβιτς. Ησυχία παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω είναι εκτίμησή μου για τη δυνατότητα που μου δίνεται να απαντήσω σε ορισμένα από τα σχόλια που έγινε. Είναι σημαντικό να είναι πάρα πολύ σωστά νομικά ρυθμισμένη αυτή η υπόθεση. Να μην ε, υπάρχει δυνατότητα προσβολής ε, από κάποιους της ε, δυνατότητας λειτουργίας της Επιτροπής μεσούσης μιας ε, ερευνητικής διαδικασίας. Πιστεύω ότι είναι προς όφελος όλων αυτό. Η κυρία Γιάτεν και άλλοι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ζήτημα της αποκάλυψης ε, εμπιστευτικών πληροφοριών. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό θα χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία για να βρούμε μια καλή λύση και για τα τρία θεσμικά όργανα. Επίσης, ε, εκτιμώ πάρα πολύ τα σχόλια του κυρίου Χέφνερ, ο οποίος τόνισε σαφώς τη σημασία ε, των απόρριτων στοιχείων που φτάνουν στι εξεταστικέ επιτροπέ. Και επίση θα ε, αυτό που είπε ο κύριο ε, Νταφ που υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τη μη συμμεταχείριση των εθνικών δημοσίων υπαλλήλων με του Ευρωπαϊκού. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το πνεύμα συνεργασία και να βρούμε μια λύση που θα είναι αποδεκτή και για τα τρία θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Τελευταίο ομιλητή για να κλείσει η σημερινή συζήτηση είναι ο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο κύριο ε, Βάμεν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κύριε Επιτροπέ, θα ήθελα καταρχά να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε να συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση υψηλή ποιότητα στο Κοινοβούλιο σήμερα. Ξέρω ότι αυτό το θέμα σας είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι ότι το Συμβούλιο και η Ιδανική Προεδρία ε, σέβεται πάρα πολύ το δικαίωμα πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα. Προσβλέπω στην ψήφιση της έκθεσης Μάρτιν και πρέπει να σας πω ότι η Προεδρία μας ε, θα εξετάσει με μεγάλη επιμέλεια την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε ε, κάποια από τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων. Ε, θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που να ικανοποιούν και το Κοινοβούλιο και τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ ιδιαίτερα τον κύριο Μάρτιν για το επικοδομητικό του πνεύμα και την προθυμία εξέβρεση συμβιβασμών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Χαιρόμαστε για αυτή την ευελιξία, για αυτή την επιθυμία διαπραγμάτευσης και είμαστε πεπισμένοι ότι Στη συνεργασία με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτέ οι επιτροπές να εργάζονται όσο γίνεται καλύτερα. Αλλά θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε η Εξεταστική Επιτροπή να εργάζεται με τον τρόπο που ορίζει η συνθήκη και να σέβεται ε, το ρόλο και τι αρμοδιότητε των άλλων θεσμικών οργάνων. Με χαρά λοιπόν θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο σα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Ε, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει τη συζήτηση, ψηφοφορία ε, ακολουθεί σε λίγο στις 12 και 10. Ευχαριστώ πολύ.